Hello everyone. Hello everyone. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που καλωσορίζω την Κρέτα Θούμπεργκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θέλω να καλωσορίσω επίσης και την κυρία Τσότ, υφυπουργό εκπρόσωπο της Ζουρμανικής Προεδρίας, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι εδώ, να τονίσω την παρουσία της κυρίας Κοράτσα Μίλ, που είναι συντονίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την τελευταία μας ολομέλεια και την τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος πριν τις εκλογές του Μαΐου. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κλείσει με καλύτερο τρόπο τις εργασίες μας παρά με την παρουσία εδώ μιας τόσο νέας υποστηρίκτριας ε, του κλίματος όπως η Γκρέτα. Δεν χρειάζεται να κάνω λεπτομερής, ε, λεπτομερής αγωγή της Γκρέτα. Την ξέρουν όλοι σε πολλά επίπεδα. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την για την ε, μόνιμη και χωρίς εμπόδια δέσμευσή της προς όφελος Τη μάχης κατά της αλλαγής του κλίματος και να την ευχαριστήσω που δέχθηκε να έρθει στο Κοινοβούλιο ε, και να μοιραστεί μαζί μας ε, τις απόψεις της για ένα θέμα που είναι από τα πιο σημαντικά θέματα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις ευρωεκλογέ. Η Γκρέτα ταξίδεψε μεγάλη απόσταση με τρένο από την Σουηδία κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών της για να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του, των των πεπιθήσεών της και της δέσμευσης που έχει αναλάβει. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, δεν μιλάμε μόνο, βλέπουμε τις, την πρακτική συνέπεια του να εμπλέκονται όλοι οι φορείς όλων των ηλικιών και από κάθε επίπεδο της κοινωνίας στην ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ξέρουμε ποια είναι η δουλειά μας. Ήμασταν υπερβολικά φιλόδοξοι, ίσως το πιο φιλόδοξο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας στόχους του κλίματος για την Ευρώπη στα επόμενα έτη. Ξέρουμε ότι η φιλοδοξία αυτή πρέπει να υποστηριχθεί και να συνεχιστεί και από την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν θα πω περισσότερα, Ήδη έχουμε μια μικρή καθυστέρηση και ξέρω πως όλοι περιμένετε να ακούσετε τις απόψεις της Γκρέτα. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να μιλήσετε. Καθιστή ή όθια προτιμάτε να μιλήσετε, όπως προτιμάτε. Okay. Κοντά στο μικρόφωνο, αν γίνεται, να μιλάτε. So, <laughs> you see, you're a bit far from it. Yeah. But we will make it quiet, so we'll hear you. Θα, έχουμε, θα κάνουμε ησυχία μέσα στην αίθουσα, οπότε θα ακούγεσαι. Name... <laughs> I'm sorry. My name is... Ονομάζομαι Κρέντα Τούνμπεργκ. Είμαι 16 χρονών Είμαι από τη Σουηδία και θέλω να πανικοβληθείτε. Θέλω να κάνετε σαν να έχει πάρει φωτιά το σπίτι σας. Αυτά τα λόγια τα έχω ξαναπεί. Και πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει και μου έχουν εξηγήσει γιατί είναι μια κακή ιδέα αυτό. Πάρα πολλοί πολιτικοί μου έχουν πει και μου έχουν εξηγήσει ότι ο πανικός ποτέ δεν οδηγεί σε τίποτα το θετικό. Και συμφωνώ. Συμφωνώ ότι αν πανικοβάλλεσαι ε, χωρίς πραγματικά να χρειάζεται είναι πολύ κακή ιδέα. Όμως, όταν έχει πιάσει φωτιά το σπίτι σου και θέλεις το σπίτι σου να το κρατήσεις, να μην καταδαφιστεί από τη φωτιά, τότε ένας βαθμός πανικού χρειάζεται. Ο πολιτισμός μας είναι εύθραυστος. Είναι σαν ένα κάστρο στην άμμο. Η πρόσωψη είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα θεμέλια Κάθε άλλο παρά γερά είναι. Έχουμε κόψει τόσες πολλές γωνίες. Χτες ο κόσμος με απόγνωση και τεράστια θλίψη παρακολουθούσε πώς κατέρεε τμήμα της Παναγίας των Παρισίων. Κάποια κτίρια δεν είναι μόνο κτίρια, αλλά θα ξαναχτιστεί η Παναγία των Παρισίων. Ελπίζω τα θεμέλια της να είναι γερά Ελπίζω τα δικά μας τα θεμέλια να είναι επίσης γερά. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι. Γύρω στα 2030, 10 χρόνια, 259 ημέρες και 10 ώρες από τώρα, θα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου θα έχουμε μια μη αναστρέψιμη αλυσιδωτή αντίδραση εκτός ελέγχου που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει και στην καταστροφή του πολιτισμού μας. Εκτός, εκτός αν μέχρι τότε γίνουν αλλαγές, μόνιμες αλλαγές χωρίς προηγούμενο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, τουλάχιστον κατά 50%. Και σημειώστε παρακαλώ ότι αυτοί οι υπολογισμοί δεν... Ε, μάλλον ότι αυτοί οι υπολογισμοί εξαρτώνται και από εφευρέσεις που δεν έχουν καν γίνει ακόμα, που μένει να γίνουν. Εφευρέσεις, τεχνολογία δηλαδή, που θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα από, αυτά τα, τις, από αυτές τις αστρονομικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα που έχουν σήμερα. Επιπλέον οι υπολογισμοί αυτοί δεν προβλέπουν και απρόβλεπτα όπως ε, για παράδειγμα το μεθάνιο, το οποίο βγαίνει από το πέρμαφρόστ στην Αρκτική. Ούτε λαμβάνουν υπόψη την συνεχή θέρμανση του πλανήτη εξαιτία της ε, ρήπανσης του αέρα. Ούτε μιλάμε για δικαιοσύνη, για κλιματική δικαιοσύνη, ε, πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στη Συμφωνία των Παρισίων και που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να πετύχουμε τις αλλαγές που θέλουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι πρόκειται για υπολογισμούς, πρόκειται για εκτιμήσεις, δηλαδή ότι τα σημεία αυτά χωρίς επιστροφή μπορεί να προκύψουν πολύ νωρίτερα από το 2030. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος και να το πει με βεβαιότητα. Όμως, είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα συμβούν αυτές οι καταστροφές μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια λίγο πολύ. Γιατί οι υπολογισμοί αυτοί δεν είναι απόψει γνώμης, ε, δεν είναι πράγματα που μαντεύουμε. Βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα τα, στα οποία έχουν καταλήξει όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο IPCC. Και γι' αυτό και εμείς στηρίζουμε το έργο του IPCC, παρόλο που δεν το στηρίζουν όλοι. Εμείς Βρισκόμαστε στα μέσα σήμερα της έκτης μασικής εξαφάνισης και η εξαφάνιση των ειδών σήμερα συμβαίνει 10.000 φορές πιο γρήγορα από ό,τι κανονικά. Κάπου 200 είδη εξαφανίζονται κάθε μέρα από τον πλανήτη μας. Η διάβρωση γόνιμων εδαφών, η καταστροφή των δασών μας, η τοξικότητα στον αέρα μας, το ότι χάνεται η ζωή άγριων ειδών, εντόμων, ότι οι ωκεανοί μας γίνονται περισσότερο όξινοι. Όλα αυτά είναι καταστροφές οι οποίες επιταχύνονται συνεχώς με τον τρόπο που εμείς ζούμε, με το οικονομικό μοντέλο που ακολουθούμε εμείς εδώ σε αυτό το κομμάτι του κόσμου που είναι τόσο τυχερό να μπορεί να απολαύσει αυτή την οικονομική ευημερία. Σχεδόν όμως κανείς δεν γνωρίζει για αυτές τις καταστροφές ή καταλαβαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μόνο τα πρώτα λίγα συμπτώματα αυτής της κλιματικής και οικολογικής καταστροφής. Και είναι λογικό, κανείς δεν τους τα έχει πει ή ακόμα πιο σημαντικό, δεν τους τα έχει πει ο σωστός άνθρωπος και με το σωστό τρόπο. Το σπίτι μας λοιπόν γκρεμίζεται και οι ηγέτες μας πρέπει να αρχίσουν να δρουν, γιατί δεν το κάνουν αυτή τη στιγμή. Αν το σπίτι μας καταραίει, οι ηγέτε μας, οι επικεφαλείς μας δεν θα έπρεπε να συνεχίζουν όπως κάνουν σήμερα, θα έπρεπε να φροντίσουν να αλλάξουν τα πάντα στη συμπεριφορά τους, όπως όταν έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Αν ε, το σπίτι μας ε, κατέρεε, γκρεμιζόταν, τότε δεν θα ταξιδεύατε σε business class αεροπλάνα ε, λέγοντας ότι η αγορά θα τα λύσει όλα και προβλέποντας μερικές μικρές έξυπνες λύσεις σε μεμονωμένα προβλήματα. Ούτε θα προσπαθούσατε να βγείτε από την κρίση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπήκατε σε αυτή, δηλαδή καταναλώνοντας όλο και περισσότερο. Αν το σπίτι σας κατέρεε, δεν θα είχατε τρεις διασκέψεις κορυφής έκτακτες για το Brexit και καμία όσον αφορά το κλίμα ή τα οικολογικά συστήματα και το περιβάλλον. would... Ούτε θα συζητάγατε για την απάλληψη του άνθρακα σε 15 ή σε 11 χρόνια. Αν το σπίτι σας γκρεμιζόταν δεν θα γιορτάζατε το ότι μία μόνο χώρα η Ιρλανδία ίσως σύντομα αποκλείσει τα ορυκτά από τα καύσιμά της. Ούτε θα γιορτάζατε το γεγονός ότι η Νορβηγία αποφάσισε να σταματήσει τις εξορίξεις στο Λόφοτεν, αλλά αλλού θα συνεχίσει την εξόριξη πετρελαίου. Έχουμε αργήσει 30 χρόνια για τέτοιου είδους εορτασμούς. Αν το σπίτι μας γκρεμιζόταν τα μέσα ενημέρωσης μόνο γι' αυτό θα γράφαν, τίποτα άλλο. Θα ήταν πάντα στους τίτλους η κλιματική και οικολογική κρίση την οποία διανύουμε. Αν το σπίτι μας γκρεμιζόταν, δεν θα λέγατε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και θα βάζατε στα χέρια εφευρετών και τεχνολογικής προόδους μόνο την ε, κατάσταση και τις ζωές ε, των ειδών και των ανθρώπων. Ούτε οι πολιτικοί θα συζητούσαν τόσο πολύ για φόρους και Brexit. Αν πραγματικά τρέμανε οι τύχοι του σπιτιού μας και γκρεμιζόντουσαν, τότε σίγουρα θα βάζατε τις διαφορές σας στην πάντα και θα συντονίζατε τη δράση σας, συμφωνώντας για κάτι. Well, ε, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι το σπίτι μας γκρεμίζεται. Και δεν έχουμε πια χρόνο. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν συμβαίνει ουσιαστικά. Ο καθένας και τα πάντα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί λοιπόν να σπαταλάμε τόσο πολύτιμο χρόνο συζητώντας για το ποιος πρέπει πρώτα να κάνει τις αλλαγές αυτές. Όλοι και όλα πρέπει να αλλάξουν αλλά όσο πιο μεγάλο είναι το βήμα στο οποίο βρισκόσαστε, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχετε. Τόσο, όσο πιο μεγάλο είναι το αποτύπωμά σα άνθρακα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ηθική σα ευθύνη και καθήκον. Λοιπόν, λέω στου πολιτικού ότι τώρα πρέπει να δράσουν. Όταν του το λέω όμω, τι μου λένε, είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα δραστικό γιατί δεν θα είναι δημοφιλέ στου ψηφοφόρου του. Και έχουν δίκιο γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν γιατί χρειάζονται αυτές οι αλλαγές, γιατί απαιτούνται. Και γι' αυτό εγώ συνεχίζω να σας λέω να ενωθείτε πίσω από τους επιστήμονες, να ακούσετε τι λένε οι επιστήμονες και να βάλετε την επιστήμη στην καρδιά της πολιτικής και της δημοκρατίας. Έχουμε εκλογέ ε, σύντομα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί, πολλοί από εμά που μα επηρέαζε ακόμα περισσότερο η κρίση αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμένα, δεν μπορούμε καν να ψηφίσουμε ούτε είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε τις ε, αποφάσεις που διαμορφώνουν οι επιχειρήσεις, η πολιτική, τα μέσα ενημέρωση, εκπαίδευση κτλ. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και εμείς τις αποφάσεις και δεν υπάρχει χρόνος. Και γι' αυτό και εκατομμύρια παιδιά βγαίνουν στους δρόμους, απεργούν για το κλίμα, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος την κρίση αυτή για το κλίμα. Πρέπει να μας ακούσετε εμάς που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Πρέπει εσείς να ψηφίσετε για μας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν μπορεί να ξεγίνει αργότερα. Με τις εκλογές αυτές ψηφίζετε για τις μελλοντικέ συνθήκες ζωής του ανθρώπινου είδους. Και παρόλο που οι πολιτικοί που χρειάζεται σήμερα, οι πολιτικοί μάλλον που χρειάζονται σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν εναλλακτικέ και διάβασα σε εφημερίδες ότι κάποια κόμματα δεν με θέλουν καν σε αυτό το βήμα, γιατί δεν θέλουν να συζητιέται το θέμα του κλίματο. Το σπίτι μας γκρεμίζεται λοιπόν. Το μέλλον και ό,τι έχουμε κερδίσει από το παρελθόν είναι στα χέρια μας σήμερα. Δεν είναι ακόμα πολύ αργά για να δράσουμε. Χρειάζεται βέβαια μεγάλο όραμα, χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται αποφασιστικότητα για να δράσουμε τώρα, για να φτιάξουμε τα θεμέλια πολύ πριν αρχίσουμε να μιλάμε για το ταβάνι. Δηλαδή χρειάζεται να σκεφτούμε όπως όταν φτιάχνουμε ένα καθεδρικό. Σας παρακαλώ λοιπόν ξυπνήστε και κάντε τις αλλαγές που απαιτούνται. Κάντε ό,τι μπορείτε. Αλλά ακόμα και αυτό δεν φτάνει, γιατί όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ωραία, μπορεί να μην θέλετε να μ' ακούτε. Στο κάτω-κάτω δεν είμαι παρά μια μαθήτρια 16 χρονών από τη Σουηδία. Όμως δεν μπορείτε να γνωρίτε τους επιστήμονες. Ούτε την επιστήμη, ούτε τα εκατομμύρια μαθητές που απεργούν για το δικαίωμά τους στο μέλλον, για το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον. Σας παρακαλώ, μην αποτύχετε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μεγκρέτα, για τις ε, κουβέντε σου, για τα λόγια σας που μας ε, ενθαρρύνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που σας ακούμε και βρίσκουμε ότι πραγματικά μας εμπνέουν τα λόγια σου. Εμπνέουν μικρού ε, μικρούς και μεγάλους. Όλους τους ανθρώπους, γενικά και τους πολιτικούς όλους ιδιαίτερους. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ζητήσω από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να πάρουν το λάγο για να μας απευθύνουν τις σκέψεις τους για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια. Γι' αυτό παρακαλώ να μην υπερβείτε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Και πρώτος είναι ο Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και σαν Αγκρέτα για την επίσκεψή σου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά μας εμπνέει ο λόγος σου. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμπνέεις και εκατοντάδες χιλιάδες νεαρούς ανθρώπους που πλέον μας ε, σπρώχνουν να κάνουμε πιο πολλά για το περιβάλλον. Και συναντήθηκα με πολλούς εξ αυτών στη δική μου επικράτεια και με εντυπωσίασε ο 14χρονος Πόλο, ο οποίος επί τρία χρόνια ήδη στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον ακτιβισμό κατά της αλλαγής του κλίματος. Νομίζω ότι και εσύ και ο Πολ και όλοι οι υπόλοιποι δεν ε, αξίζουν, δεν τους αξίζουν αυτές οι προσβλητικές κουβέντες που ακούμε κυρίως από πιο ηλικιωμένου. Τους αξίζει η υποστήριξή μας άμας. Ναι βεβαίως, χειροκροτήστε λέει ο κ. Λίζα. Και φυσικά γίνεται αυτή η μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να χάνεται ώρα σχολείου ή όχι. Εγώ τις ώρες σχολείου ακόμα και από τους δασκάλους μου ε, με παράτρενα να βγω στους δρόμους και να διαδηλώσω για το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Γερμανία. Και συμφωνώ λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτό, φυσικά να γίνεται εκτός όρων σχολείου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η αλλαγή του κλίματος. Και η αλλαγή του κλίματος κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί η μεγαλύτερη πρόκληση για την πολιτική μας γενιά. Και αυτά δεν είναι δικιά μου λόγια, δεν είναι τα λόγια του Μάνφρετ Βέμπερ, ο οποίος ε, επικύρωσε τη συνθήκη του Παρισιού. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και πολλά παραπάνω. Ακόμα και αν πολλές φορές δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη μπορεί να μην κάνουν αρκετά πράγματα, αλλά είναι σημαντικό γιατί χωρίς την Ευρώπη δεν θα είχαμε καν τη Συμφωνία του Παρισιού. Και γι' αυτό λοιπόν αυτές είναι οι κουβέντες του Τόπστερν ε, του πρώην Συμβούλου του Μπαράκ Ομπάμα, που ήταν ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δήλωσε ότι χωρί την Ευρώπη δεν θα ήμασταν πουθενά, δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα. Αλλά να μα πρόξετε λοιπόν να πετύχουμε πιο παραπάνω πράγματα. Χωρί την Ευρώπη δεν θα είχαμε πετύχει καν αυτά τα λίγα που έχουμε πετύχει. Για το μέλλον έχουμε δύο σημαντικά θέματα και ελπίζω και εσεί και οι νεαροί που σκέφτονται όπω εσύ να συμφωνούν. Θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι προ το περιβάλλον έχει κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έχει υποστηρίξει τα κράτη-μέλη. Δεν είναι όμω ε, το Κοινοβούλιο, συγγνώμη, δεν την έχουν υποστηρίξει ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να σπρώξουμε λοιπόν, να παροτρύνουμε του αρχηγού κρατών να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Και θα πρέπει να γίνει αυτό τώρα, όχι του χρόνου. Δεύτερο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ. Α, με απασχολεί όλο ο συχνά στην επικράτειά μου έρχονται και μου μιλάνε κάθε εβδομάδα νεαρά παιδιά από το σχολείο. Γιατί η αεροπορία δεν βοηθά το κλίμα. Είναι άδικο, είναι εντελώς άδικο όταν παίρνει κανείς ε, το τρένο, το λεωφορείο, πληρώνει πολλούς φόρους, πολλά τέλη και όταν παίρνει κανείς το αεροπλάνο η αεροπορία συμμετέχει μόνο 15% ε, ε, στο σύστημα εμπορίας ρήπων. Μόνο 85% είναι δωρεάν. Αλλά ακόμα και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο υπάρχουν άτομα τα οποία πιστεύουν ότι ακόμα και αυτό το 15% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να πετύχουμε κάτι παραπάνω νομίζω. Δεν μπορούμε με τις τρέχουσες συνθήκες να απορρίψουμε ακόμα και τις ευθύνε που έχει αναλάβει η αεροπορία. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να συνεργαστούμε με τους νέους για να τα πετύχουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Ο επόμενος. Ο μιλητής, η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Γκρέτα, που ήρθε εδώ. Εκπροσωπώ του σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είμαι όμως εδώ και ω μητέρα δύο παιδιών, ενός πεντάχρονου και ενός δίχρονου παιδιού. Όταν μας μίλησες και μας έδινες τις ανησυχίες που έχουν άτομα της ηλικία σου και νεότεροι, πρέπει να πω ότι αισθάνομαι τι ίδιε τύψει που δημιουργείς και εσύ γύρω σου βλέπεις ένα άτομο, ε, βλέπεις άτομα στην αίθουσα που χειροκροτούν αυτά που λες, αλλά στο τέλος τα ίδια πάντα συμβαίνουν. Όταν μπαίνουμε στην ουσία, όταν φτάνουμε στην νομοθεσία που μπορούμε να υιοθετήσουμε, καταλήγουμε να μειώνουμε τις φιλοδοξίες μας. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν και πιστεύω ότι και η εμπειρία των συναδέλφων το ίδιο δείχνει. Δεν είναι η πρώτη φορά όταν μιλάμε για πραγματικά νομοθετικά κείμενα, στην ουσία κάνουμε πίσω ή παναχωρούμε λόγω πιέσεων από τα διάφορα λόμπι. Το λέω αυτό έχοντας παλέψει για τη μείωση των εκπομπών και στα επιβατικά αεροσκάφη και στα οχήματα, αλλά το ίδιο συμβαίνει παντού, θα σας το πούν όλοι οι συνάδελφοι. Είσαι μία απλή 16χρονη ε, μαθήτρια. Εγώ έχω την Μάλτα, το μικρότερο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα όμως δεν είναι ούτε ηλικία ούτε προέλευση, αλλά είναι ε, θέμα αποφασιστικότητας να προχωρήσεις, να πιέσεις για τις αλλαγές. Από αυτά που είδα όταν σε άκουγα πριν και σήμερα, θεωρώ ότι έχει την αποφασιστικότητα και επηρεάζει αυτή η αποφασιστικότητα και άλλους, όχι μόνο νέους και μεγαλύτερους. Έχω δει νέους να βγαίνουν στους δρόμους, ακόμα και στη χώρα μου, φωνάζοντας, προσπαθώντας να περάσουν τη φωνή τους ό,τι αφορά την αδράνεια για το κλίμα. Λε, είπε μάλλον ότι ω 16χρονοι δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Κάποια κράτη-μέλη επιτρέπουν σε 16χρονου να ψηφίσουν και νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση σε αυτό. Η Μάλτα, η Αυστρία επιτρέπουν την ψήφο των 16χρονων. Το θέμα δεν είναι θέμα αποφάσεων ανάλογα με την ηλικία του καθενός. Οι αποφάσεις στις εκλογές αυτές επηρεάζουν τους 16χρονους και που σε 5 χρόνια θα είναι 21 ετών. Εσείς θα υποστείτε τις επιπτώσεις των, απο... αποφάσεων που λαμβάνονται σήμερα. Και θεωρώ ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να πιέσουμε ώστε οι νέοι να έχουν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και χαίρο που ανέφερε ο συνάδελφος ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μπροστά μας είναι η αλλαγή του κλίματος. Όντως αυτό είναι και χρειάζεται δράση. Και αν θέλετε, μακριά από τις κάμερες, θα ήθελα όλοι να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και δράση. Γιατί αν δεν ενδιαφερθούμε για τον πλανήτη μας δεν θα έχουμε ούτε οικονομίες ούτε δουλειές να φροντίσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται και βγάζουν μεγάλους λόγους αλλά δεν τους υλοποιούν. Μίλησε ο συνάδελφος για διάφορους συναδέλφους. Εγώ θέλω να κλείσω με μια παράθεση δική σου πριν από λίγο καιρό που με εντυπωσίασε. Είπες ότι πρέπει να ότι έχουμε υπόλογες γενναίες. Δεν μπορούμε, πρέπει να οργιστούμε και αυτή την οργή να τη μετατρέψουμε σε δράση. Αυτό χρειάζεται για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα μιλήσω στην μετρική μου γλώσσα, αν μου επιτρέπετε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά. Eh, εγώ εκπροσωπώ εδώ την ομάδα του ECR και εγώ είμαι και πατέρας και παππούς και σας καλωσορίζω και εξ ονόματος της δικής μας ομάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να πω ότι κινήσατε πολλά πράγματα, χιλιάδες νέους οι οποίοι ενθουσιοδός ε, δραστηριοποιούνται για να προωθήσουμε την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και στη δική μου την πατρίδα, στη Φλάντρα, βγαίνει ο κόσμο βγαίνουν οι νέοι κατά χιλιάδες στου δρόμου και σα ε, υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά τώρα που φαίνεται που δεν πάτε στο σχολείο λιγότερο. Αυτό που μα απασχολεί λοιπόν είναι το περιβάλλον μας και ξεκινάμε λοιπόν μια δράση που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια και φυσικά είμαστε περιορισμένοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα τελευταία πέντε χρόνια εργάζομαι για τη βιοπικιλότητα, για μια κυκλική οικονομία και για την υπεύθυνη ε, διαχείριση των πλαστικών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε πετύχει πολλά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα μεγάλο νομοθετικό πακέτο έχει ολοκληρωθεί και αυτή την εβδομάδα θα ψηφίσουμε την πρώτα πρότυπα του του άνθρακα για τα νέα φορτηγά και το νέο πρόγραμμα LIFE για την ε, φύση και τη βιοπικιλότητα. Και αυτό που πάντα πίστευα είναι ότι η οικονομία και η οικολογία θα πρέπει να συμπληρωθούν με ρεαλισμό και με μεγάλο επίπεδο φιλοδοξίας, γιατί μόνο έτσι στον πραγματικό κόσμο πετυχαίνουμε πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν το κόμμα μου θέλει να ε, προωθήσει την οικολογική μετάβαση στα πλαίσια της προόδου και της ανάπτυξης, γιατί θα πρέπει πολιτική μας όχι μόνο να προστατεύσει την οικολογία και το περιβάλλον, αλλά και τις θέσεις εργασίας. Άρα χρειαζόμαστε πραγματική καινοτομία και δημιουργικότητα. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδί και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και είμαι απόλυτα πεπισμένο. και γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε τους νέους μας για να βρούμε πιο πολλές λύσεις, για να πετύχουμε τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν πραγματικά με λυπεί αυτή η τοπάθεια, η εντύπωση ότι δεν θα υπάρχει μέλλον, γιατί κάθε μέρα πολλοί κόσμος ψάχνει και βρίσκει λύσεις. Βρίσκει λύσεις που θα συμβάλλουν στην ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, παρά το γεγονός ότι, μάλλον πρόσφατα, ε, βρήκαν ε, στο Πανεπιστήμιο του Λόβεν κάποια ηλιακά πάνελ που βγάζουν ε, ενέργεια από την ατμόσφαιρα. Ένα παράδειγμα μόνο που θα λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε στις νέες τεχνολογίες μια ευκαιρία και έχω υπόψη μου για παράδειγμα την βιοτεχνολογία, την πυρηνική ενέργεια στο ε, ενεργειακό μείγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγετική δύναμη, αλλά μια παγκόσμια πρόκληση χρειάζεται παγκόσμιες ε, λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε συμμάχους και ελπίζω από βάθος καρδιάς ε, ότι οι νέοι θα αναγνωρίσουν ε, την ανάγκη για την καινοτομία και θα μπορέσουν να την υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονικό όριο για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τορβάλτ έχει το λόγο. Ναι, εγώ θα μιλήσω στην γλώσσα της Γκρέτα. Γεια σου, Γκρέτα, και καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είχε λίγο μεγαλύτερη πλάκα να με λέγανε Χάντζελ, να μην λεγόμασταν Χάντζελ και Γκρέτα, που βγήκαμε από το μεγάλο δάσο και προσπαθούμε να, κάνουμε τη ζωή δύσκολο, δύσκολη στην ε, μάγισσα της αλλαγής του κλίματος. Δυστυχώς δεν ονομάζομαι Χάνσελ, αλλά σίγουρα και από την προφορά μου ακούσω ότι είμαι από τη Φινλανδία. Έχεις έρθει λοιπόν στο σωστό μέρος, Γκρέτα. Γιατί αν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή όταν μιλάμε για το κλίμα και το περιβάλλον, είναι αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα λαμβάνουμε και τις αποφάσεις του μέλλοντος και θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε την, ε, το μέλλον το οποίο περιγράφεις. Να σας πω επίσης ότι δεν είμαι εδώ για το δικό μου λογαριασμό. Είμαι εδώ για τα εγγόνια μου. Έχω τρία εγγόνια τα οποία είναι λίγο πιο μεγάλα σε ηλικία από ότι εσύ και έχω και τρία εγγόνια λίγο πιο νεαρά. Όταν θα επιστρέψω λοιπόν στο σπίτι στη Σουηδία, στην ε, Φιλανδία, θα με ρωτήσει, μίλησε τελικά στην Κρέτα. Και τώρα λοιπόν μπορώ να απαντήσω ότι ναι. Τη μίλησα και υποσχέθηκα ότι θέλω να είμαι καλύτερο παππού και καλύτερο ε, βουλευτή. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε λάβει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων. Και κατά πάσα πιθανότητα έχει δίκιο όταν λες ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα ακόμα. Προσπαθήσαμε όμως να ρυθμίσουμε τα πράγματα με την εμπορία ρήπων, προσπαθήσαμε να λάβουμε δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και τις κατασκευές, να πετύχουμε πιο εύκολα τους στόχους που έχουμε θέσει. Λάβαμε αποφάσεις για τη χρήση της γης και επίσης αγωνιστήκαμε για τον περιορισμό των ρήπων από τα οχήματα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όμως. Όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ηλεκτρικά οχήματα στο μέλλον. Αν όμως ε, χρησιμοποιούν βρώμικη ηλεκτρική ενέργεια, ουσιαστικά ρηπαίνουν πιο πολύ από ό,τι και τα ντίζελ τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να ανανεώσουμε το σύστημα ηλεκτροδότησης και αυτό θα αποτελέσει μία από τι μεγάλε προκλήσει του μέλλοντος. Ένα πράγμα σου υπόσχομαι, Γκρέτα. Θα σε επισκεφτώ στην Σουηδία όταν θα λάβουμε τις αποφάσεις τις οποίες μας ζητάς να πάρουμε. Μπορεί να μην είναι αύριο ή μεθαύριο, μπορεί να μας πάρει κάποια χρόνια, αλλά νομίζω από ό,τι ακούς και από τα χειροκροτήματα εδώ στην αίθουσα, όλοι πιστεύουμε ότι κάνεις κάτι σωστό και θέλουμε να σε υποστηρίξουμε. Thank you very much. Ο κύριος Έικχαουτ, επόμενος Καλώς Γκρέτα. Και ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει να σε ευχαριστούν οι πολιτικοί, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί τώρα ξέρουμε ότι οι επόμενες εκλογές θα αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Σήμερα οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα πάνε στις ευρωεκλογέ γιατί ενδιαφέρονται για το κλίμα. Και αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη δουλειά που έκανε εσύ και οι άλλοι μαθητές και φοιτητές. Έρχομαι από ένα πράσινο κόμμα και θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή. Κατάφερες κάτι τέτοιο. Εμείς παλεύαμε για χρόνια χωρίς να είμαστε τόσο επιτυχημένοι όσο εσύ. Να στραφώ τώρα στους συναδέλφους. Θα μπορούσα να γίνω κοινικό, μιλώντας για το παρελθόν, τι διάφορες ψηφοφορίε που είχαμε και τις συζητήσει που κάναμε. Δεν είδα να επίγεστε τόσο όσο σήμερα στην αίθουσα, αλλά ας δούμε το μέλλον καλύτερα όντας όλοι εδώ. Τον Ιούλιο, όταν ψηφίσουμε για ένα νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί από εσά επιστρέψετε, ελπίζουμε. Εγώ ελπίζω όλα τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου που χειροκροτήσαμε σήμερα την Κρέτα θα θυμώνται ότι θα πρέπει να δουν και το πρόγραμμα του νέου Ευρω... Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δουν αν έχει αλλάξει όντως η πολιτική. Αν έχουμε αλλάξει πολιτικές για την διακοπή χρήσης του άνθρακα, για να πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, για να μην πληρώνουμε ούτε μία, ένα ευρώ επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα πολιτικές που μέχρι τώρα δεν έχουμε υλοποιήσει. Ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Ψηφίστε όμως για το πρόγραμμα αυτό του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο, γιατί μόνο τότε το χειροκρότημα θα έχει νόημα. Να στραφώ προς τον Επίτροπο. Έχετε μια ευκαιρία ακόμα κύριε Επίτροπε. Το Σεπτέμβριο θα πάτε στη Νέα Υόρκη, στη Σύνοδο Κορυφής του ΙΕ για την αλλαγή του κλίματος. Σήμερα είναι μια καλή στιγμή να υποσχεθείτε ότι θα πάτε στη Νέα Υόρκη και θα πείτε ότι η Ευρώπη θα αυξήσει τους στόχους για το κλίμα το 2000, μέχρι το 2030. Θα το κάνετε. Να πω δυο λόγια και προς την Προεδρία. Έχετε στις 9 Μαΐου τη Σύνοδο Κορυφής για το μέλλον της Ευρώπης στο Σύμπιου. Θα ε, διασφαλίζει ότι τότε το Συμβούλιο και όλα τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν το πρόγραμμα ουδετερότητας του κλίματος το 2030 έως και τη μείωση των εκπομπών μας περισσότερο ε, μέχρι τότε, μόνο τότε θα είναι επιτυχημένη η Σύνοδος Κορυφής, γιατί τότε τα λόγια θα έχουν γίνει πράξη. Και ευχαριστώ για όλα αυτά την Κρέτα Τούνμπεργκ. Thank you, Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόιλαν. Λίν Μπόιλαν λέγομαι από την αριστερά. Και θέλω πραγματικά να εκφράσω τη χαρά μου που σε βλέπω εδώ η, ωστόσο, οι εξελίξεις του τελευταίου μήνα έδειξαν τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι πολιτικές ομάδες που ήθελαν να σε εμποδίσουν να μιλήσει σήμερα είναι αυτές που αποφάσισαν κατά της, ε, α, ε, της ανάκλησης της πρόσβασης στην ExxonMobil για το κοινοβούλιο. Η Exxon έδωσε εκατομμύρια προσπαθώντας να υπονομεύσει την αλήθεια. Ξέρουμε ότι τα κεκτημένα συμφέροντα έχουν την πολιτική πλειοψηφία, έπεισαν ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος με συνεχή ανάπτυξη. Και ξέρω ότι χρησιμοποιούμε τώρα ήδη περισσότερους πόρους από ό,τι είναι βιώσιμο. Και ο Σάκη η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι το, η θερμοκρασία ανεβαίνει 3% το χρόνο. Αυτό είναι παράλογο. Δεν μπορεί η οικονομία να αντιμετωπίζεται ως χωριστό παράγοντα και όλα τα άλλα να, παρα, να μένουν ε, πίσω. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς να αντιμετωπίσουμε την οικονομία και η αλλαγή του κλίματος είναι μεγαλύτερη κρίση. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε τις επιχειρήσεις και να ενωθούμε γύρω από αυτά που λέει η επιστήμη, όπως είπε η Γκρέτα. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπε σήμερα η Γκρέτα. Ανέφερε στην Ιρλανδία, τη χώρα μου, και το πώς αλλάζει απομακρυνόμενη από τα ορυκτά καύσιμα, παρότι χορηγούνται ακόμα άδειε εξόριξη σε εταιρείε, ε, συνεχίζει να σκέφτεται την εγκατάσταση νέων τερματικών αερίου. Ε, όσοι έχουν πολιτική εντολή, έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν για να, να πολεμήσουν για μια ταχύ αντιμετώπιση του κλίματος, όχι για να νεύουν καταφατικά και να χειροκροτούν, να δρουν με βάση τις πολιτικές εντολές που έχουν λάβει για να, λάβ, αναλάβουν τα μεγάλα μέτρα που, που απαιτούνται. Δεν πρέπει να επενδύουν εκατομμύρια σε υποδομές για ορυκτά καύσιμα. Δεν πρέπει να περιορίζουν τις ε, φιλοδοξίες μας μόνο στο 0,5 βαθμούς αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να, όπως σωστά είπες, όχι μόνο να κάνουμε αγώνα κατά του, να κάνουμε συνόδους κορυφής για το Brexit, αλλά και για το κλίμα. Χρειαζόμαστε λιγότερη παραγωγή εξόριξης, μεγαλύτερη τοπικοποίηση εις βάρος της παγκοσμιοποίησης. Με άλλα λόγια, είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσγειωθεί. Σας ευχαριστώ για την έμπνευση που πέρασε σε όλους τους νέους και σε όλους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το λέω με ειλικρίνεια. Εγώ με έπεισες και με, με έκανες να αισθάνομαι ότι πρέπει να δουλέψω περισσότερο και να κάνω καλύτερα τα πράγματα όπως και όλοι μας σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ. Ο κ. για δύο λεπτά. I, I speak in Italian. So headphones. Θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ Γκρέτα και εγώ και ευχαριστώ και για τη συμβολή σου και γιατί και να ευχαριστήσω και αυτόν που ήθελε να σε φέρει εδώ για να τονίσει τη σημασία της αλλαγής του κλίματος όπως ποτέ δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Με λυπεί ωστόσο που διαπιστώνω ότι αυτό το ρόλο του συντονιστή για το κλίμα το παίρνει μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι, αντί να το κάνουμε όλοι μας να πω ένα απλό πράγμα. Πιστεύω ότι το κακό στον κόσμο δεν είναι η αλλαγή του κλίματος, αλλά το ψέμα. Πολλοί μεγάλοι, πολλοί από αυτούς και εδώ, είναι έτοιμοι να σε χειροκροτήσουν και ίσως να ξανασηκωθούν ε, για ένα standing ovation. Ουδέποτε όμως έκαναν κάτι για να εμποδίσουν το να είναι μια κοπέλα αυτή που θα ασχοληθεί με την αλλαγή του κλίματος. Για να πετύχουμε αυτό που λες εσύ, για να μπορέσουμε να παρνικοβληθούμε θα πρέπει να έχουμε ένα θάρρος που εδώ το βλέπω μόνο σε λίγους να χτυπήσουμε, να, να αγωνιστούμε κατά των πετρελαϊκών ε, εταιριών, κατά των κύριων του αυτοκινήτου, της καύσης, των απορριμμάτων και νομίζω ότι οι μάχες αυτές είναι μάχες ε, μεγάλων, ίσως λιγότερο ψεύτικες από αυτές εδώ, αλλά μεγάλων. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε την ευθύνη αυτή σε ένα κορίτσι που κανονικά θα έπρεπε να ζούσε όπως, όλα τα, όπως οι άλλες κοπέλες. Γι' αυτό ντρέπομαι πραγματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φετιτσίνη. Με κυρία Λα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως συμβαίνει συχνά, όταν γίνονται υπερβολές προς τη μία κατεύθυνση, γίνονται ε, υπερβολές και προς την αντίθετη. Έτσι λοιπόν και τώρα οι καταστροφές που έχουν γίνει και που έχουν ανεχτεί οι προηγούμενες γενιές είναι καλό να καταγγέλλονται. Αλλά μην οδηγηθούμε σε μία επικίνδυνη κατάσταση μετά από έναν αιώνα εντατική γεωργίας και υπερβιομηχανοποίησης υπέρ του κέρδους, ε, παραβλέποντας την αρχή της πρόληψης μην καταλήγουμε σε υπερβολές. Να είμαστε σοβαροί. Το να καταγγέλουμε ότι γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει και τα πάντα. Αντίθετα, επιβάλλει μέτρο. Να μιλάμε βάσει επιστημονικών δεδομένων, αξιόπιστων και να μην βασιζόμαστε σε πυροτεχνήματα που απλώς δημιουργούν αίσθηση. Πρέπει να υπάρχουν αγνές προθέσεις και αγνά λόγια χωρίς καμία πρόθεση μακριά από τα λόμπι, μακριά από τις βιομηχανίες και τις οικονομικές δυνάμεις. Μόνο η αριστεία. Αλλιώς κινδυνεύουμε να είμαστε γελοί και αντιπαραγωγικοί. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την ε, τρύπα του όζοντος και για το στρώμα του όζοντος που έχουν ε, καταρριφθεί ξανά και ξανά. Η στερία που συνοδεύει το διοξίδιο του άνθρακα, τις δραστηριότητες ε, του ανθρώπου ή των ζώων δεν χρειάζονται. Η τελευταία έκθεση του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου για την Αγρονομία όσον αφορά ε, τον άνθρακα και τη γεωργία δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν σωστοί υπολογισμοί και αξιόπιστοι. Ναι, φυσικά και πρέπει ο άνθρωπος να σταματήσει να υπερβάλλει και ανεξέλεγκτα να έχει αέρια του θερμοκηπίου. Χρειάζεται καινοτομία, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις οικονομικές ισορροπίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση. Όλα να γίνονται με καθαρό πνεύμα και με μέτρο. Και γι' αυτό βασιζόμαστε στη δικιά σας γενιά, δεσποινής μου. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται ο γύρος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Και τώρα την κυρία Τσότ εκ μέρους της Ρουμανικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Ε, θα φιλοξενήσει βέβαια τη διάσκεψη κορυφής του Σύπιους, οπότε εκεί θα συνεισφέρει ακόμα περισσότερο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου κάλεσε την Ρουμανική Προεδρία στην συνεδρίαση αυτή και καταρχάς θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να χαιρετήσω την ε, κυρία Γκρέτα Τάμπερκ για την δέσμευσή της στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και που μας ευαισθητοποιεί για ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους και την ευθύνη που έχουμε και φέρουμε για τον πλανήτη μας και για τους πολίτες μας, ιδιαίτερα για τις μελλοντικέ γενιές. πέρα από το ότι ξεκίνησε ένα κίνημα και αποτέλεσε πηγή έμπνευση για μία ολόκληρη γενιά. Ξυπνάτε την ε, συνείδηση των ε, παλαιότερων γενιών, των ε, γονέων, των πολιτικών, των δασκάλων, των πολιτικών ηθινόντων σε όλο τον κόσμο. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε την κλίμακα και το κατεπήγον των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Όλοι ζούμε και είμαστε μάρτυρες των καταστροφικών συνεπειών στην αλλαγή του κλίματος σε όλον τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, όπως σωστά είπε η Γκρέτα και μάλιστα σε πολλές ε, περιστάσεις, η αναστροπή και η αναστροφή και οι προσπάθειε μας για την αναστροφή του τάσεων ε, είναι ανεπαρκή. Και αυτό το επιβεβαιώνει και η ειδική έκθεση του IBCC, η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου αν δεν εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αλλαγή του κλίματος, η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά δύο βαθμούς μετά το 2060 και θα συνεχίσει να ανεβαίνει στη συνέχεια. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες αντιδράσεις σε ό,τι αφορά την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να ξεκινήσει παγκόσμια δράση και να είναι ηγετική δύναμη. Τον προηγούμενο μήνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επανέλαβαν τη δέσμευσή τους σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την, ε, το τρέχον ε, φιλόδοξο πλαίσιο νομοθεσίας εξακολουθεί να είναι ηγετική δύναμη σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος και θέλει να πετύχει τους στόχους ε, του 2000, ε, για το 2020 για την ε, αέρια θερμοκηπίου και σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, έχει α, συμφωνήσει για περαιτέρω φιλοδόξου στόχου για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και οι στόχοι αυτοί πλέον μεταφράζονται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλος ιδιαίτερος αυτοί οι νόμοι θα εξασφαλίσουν περαιτέρω μείωση των εκπομπών στη βιομηχανία, στην ενέργεια και φιλόδοξου στόχου για τα εθνικά κράτη-μέλη, για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και στου υπόλοιπου τομεί, όπω είναι τα κτίρια, οικοδομέ, μεταφορέ και τα απορρίμματα, τα απόβλητα. Αυτό σε συνδυασμό και με άλλε τομεακέ πολιτικέ, σε σχέση για παράδειγμα με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, τι προδιαγραφέ ενεργειακή προδιαγραφές και το θέμα της εκπομπής της του άνθρακα από τα οχήματα. Όλα αυτά μαζί εγγυώνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τους στόχους για το 2030 για τη μείωση των αρίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με τα δεκαετία του 90. Και επίσης να πετύχει και τους εθνικούς στόχους και τις εθνικές δεσμεύσεις για την συνθήκη του Παρισιού. Με την ευρωπαϊκή λοιπόν στρατηγική, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά στην παρούσα φάση μία ανακοίνωση την οποία θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει διάφορα σενάρια για την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών. Αυτά λοιπόν τα σενάρια θα μα βοηθήσουν να πετύχουμε μείωση του αερίου του των αερίων των θερμοκηπίων σε 100% επίπεδο μέχρι το 2050 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση συζητά λοιπόν, ε, είναι αντικείμενο ε, συζήτηση ε, στου κόλπου του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Προεδρία, η Ρουμανική Προεδρία, θέλει να συνεχιστεί η συζήτηση για όλους τους τομείς. Περιβάλλον, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, ανταγωνιστικότητα, γεωργία και χρηματοοικονομικός κλάδος. Αυτή η υπουργική συζήτηση ω τώρα έχει υπογραμμίσει το γεγονό ότι υπάρχει σωστή αναγνώριση τη ανάγκης για ανάληψη δράση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση έχει δώσει έμφαση στη σημασία να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για να πετύχουμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί στη συνθήκη του Παρισιού. Το να κινηθούμε σε μία κατεύθυνση μιας χαμηλής, ε, χαμηλού άνθρακα οικονομίας θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά για να πετύχουμε την ε, μετάβαση με κοινωνικά ισορροπημένο τρόπο για όλους. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει λοιπόν να κάνει συζητήσεις για αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα και επίσης προσβλέπουμε στις εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, σε παγκόσμιο επίπεδο στο 2019 που θα αποτελέσουν μια ευκαιρία να κινητοποιηθεί η πολιτική βούληση για να αυξηθούν οι παγκόσμιες φιλοδοξίες, όπως για παράδειγμα η Σύνοδος του Σεπτεμβρίου στο ICCC. Και αυτό λοιπόν με οδηγεί στο τέλος ε, της παρέμβασής μου. Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την διοργάνωση της σημερινής συζήτησης και θα ήθελα να κλείσω με ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ προς την Κρέτα, γιατί αποτελεί πηγή έμπνευση και γιατί διαδίδει το μήνυμα για την αλλαγή του κλίματος. Βοήθησε επίσης να βρουν φωνή οι ανησυχίε των νέων. Κινητοποιώντας ε, τις απεργιακές αυτές, τις ε, κινητοποιήσεις αυτές των ε, μαθητών για το περιβάλλον. Πιστεύω ότι και ελπίζω αυτές οι κινητοποιήσεις να, καθιστούν, να καταστούν περιττές όσο θα δώσουμε, θα δίνουμε σωστέ απαντήσεις στην αλλαγή του κλίματος για να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμού στόχου τη συμφωνία του Παρισιού. Η Ευρώπη και ο κόσμος θα χρειαστούν έξυπνους και καλά εκπαιδευμένους νεαρούς ανθρώπους για ένα μέλλον ουδέτερο προς το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. thank you for your... Ευχαριστούμε πολύ για τη δέσμευσή σας και για την αναγνώρισή σας. Ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτη τώρα. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πρώτα απ' όλα σε αυτή τη συνάντηση με την Κρέτα Τούμπερκ. Εσείς είσαστε επίτροπος ο αρμόδιος για να προωθεί αποφασιστική σημασία νομοθεσία για να καταπολεμιστεί η κλιματική αλλαγή. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κρέτα Τούμπερκ όχι μόνο που ήρθε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω επειδή έχει δώσει πρόσωπο και φωνή στους νέους, όλο και περισσότερους που αναλαμβάνουν δράση για την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και καλά κάνουν, γιατί επίγει το θέμα. Μας ζητάει να δράσουμε και πολύ σωστά το ζητάει γιατί όταν θα βρεθεί δικιά της η γενιά στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στην απασχόληση γενικά, θα είναι πολύ αργά να αλλάξουμε και να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Σε ακούμε προσεκτικά. Το μήνυμά σου μας ενθαρρύνει να κάνουμε περισσότερα και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Εμείς έχουμε ανελάβει γετικό ρόλο ως Ευρώπη. Έχουμε δράσει, συνεχίζουμε τη δράση μας, αλλά τώρα πρέπει να δράσουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο γρήγορα. Έχουμε βασίσει τη δράση μας στις τελευταίες επιστημονικές ε, ενδείξεις, στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και έτσι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα συνολικά προβλήματα. Έχουμε την Συμφωνία των Παρισίων τώρα, που σημαίνει μια ε, πολυμερής συμφωνία προκειμένου να μην επιτρέψουμε να αυξηθεί πάνω από δύο βαθμούς η θερμοκρασία, αντίθετα να μείνει στον 1,5 βαθμό. Η προσπάθεια, μάλλον το γεγονός αυτό χρειάστηκε πάρα πολλές προσπάθειες η συμφωνία αυτή. 1,5 βαθμό σημαίνει ότι χρειάζονται πολλές προσαρμογές. Ελπίζω να το αναγνωρίσει ο κόσμος. Δύο βαθμοί είναι κάτι διαφορετικό. Σημαίνει διαφορετικό κόσμο και πολύ περισσότερες δυσκολίες. Σημαίνει ότι θα ζούμε σε έναν κόσμο που δεν θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Το IPCC, η έκθεση αυτή δηλαδή του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ, μας δείχνει το δρόμο. Μας λέει πόσο μεγάλη είναι η απειλή. Μας εξηγεί όμως επίσης ότι ακόμα μπορούμε να τα καταφέρουμε αν περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς και ακόμα καλύτερα στον 1,5 βαθμό. Οι επιστήμονες το φωνάζουν ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Οι άνθρωποι το ξέρουν ότι όταν φτάσουμε στο 2050 η αύξηση της θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να συνεχιστεί καθόλου. Πόσο μάλλον το 2060-2080. Και για να καταφέρουμε να μείνουμε στο μηδέν αύξηση, πρέπει να δράσουμε πολύ νωρίτερα. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, αναλαμβάνουμε ήδη δράση η, την νομοθεσία, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ότι πρέπει να έχουμε πετύχει μέχρι το 2030 και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πριν από το 2005 να έχουμε ε, μηδέν και κάτω άνθρακα, αποτύπωμα άνθρακα και ακούμε τους επιστήμονες η κινητοποίησή μας θα συνεχίσει και η δικιά σας η κινητοποίηση θα στηρίζει τη δικιά μας δράση. Και χαίρομαι πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την κλιματική ουδετερότητα για το 2050. Και περιμένω το ίδιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν θα συζητήσει τον Ιούνιο του 2019. Ναι, μπορείτε να είσαστε σίγουρος κύριε Eckhout ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Η συζήτηση αυτή όμως πρέπει να γίνεται παντού και όχι μόνο στα δικά μας θεσμικά όργανα. Γιατί το οικονομικό μας σύστημα απαιτεί δημοκρατική συμμετοχή. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί έχει σημασία για τους Ευρωπαίους. Και όπως είπε ο κύριος Σέικχαουτ, μια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε σήμερα δείχνει ότι αυτοί που σκοπεύουν να ψηφίσουν λένε ότι το κλίμα είναι αποφασιστική σημασία για να αποφασίσουν για ποιον θα ψηφίσουν. Οι εκλογές αυτές λοιπόν δίνουν την ευκαιρία στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διαλέξουν, να βάλουν το κλίμα στο κέντρο της προεκλογικής τους εκστρατείας και να εξηγήσουν στους πολίτες και στις νέες γενιές τι έχουμε ήδη καταφέρει και τι ακόμα πρέπει να κάνουμε. Επίγει η Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι χώρες μέλη, η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις να συμφωνήσουν το στόχο αυτό της κλιματικής ουδετερότητας. Επίγει, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε 30 χρόνια μπροστά μας για να το πετύχουμε, αλλά πρέπει τις δράσεις μας να τις εκπονήσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια και να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις για να υλοποιηθεί η αλλαγή αυτή. Έχουμε φιλοδοξίες για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Έχουμε κάνει αλλαγέ στην αγορά μας, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Οι στόχοι αυτοί, οι υποχρεώσει αυτές πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο. Το 2050 να υπάρχει κλιματική ουδετερότητα, όπω είπαμε, και να βρούμε και το σωστό ρυθμό για τις αλλαγέ, που να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορε. Συγχρόνω όμω, να προστατεύσουμε και τι προποθέσει και τι συνθήκε για την ευημερία των πολιτών μας και για δικαιοσύνη. Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι εφικτά και τα δύο. Θα τα καταφέρουμε. Θα προσφέρουμε στις χώρες ένα καλό μοντέλο χωρίς να θυσιάσουμε την ευημερία και την ανάπτυξη. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα που έχει δύο όψεις όπως έχουν όλα. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε και άλλα πράγματα. Τον πόλεμο, την πείνα, το μήνυμά μου σε εσά σήμερα είναι συνεχίστε την πίεση, συνεχίστε να υψώνετε τη φωνή σας υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Πιέζετε τους πολιτικούς και όσου παίρνουν αποφάσει παντού στον κόσμο. Εμείς στην Ευρώπη θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται για να υλοποιηθεί η κλιματική ουδετερότητα. Πρόκειται για το μέλλον μα και κυρίω πρόκειται για το μέλλον σα, εσά των παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας εδώ στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θεαματικό τέλος και σωστό για να κλείσουμε μια πολύ σημαντική δουλειά που κάναμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας στο Κοινοβούλιο. Θα σας δω στην επόμενη θητεία με νέα δύναμη για να αντιμετωπίσουμε την υποβάθμιση του κλίματος και με τη βοήθεια πολλών νέων. Ευχαριστώ Γκρέτα για την παρουσία σου εδώ και καλή τύχη στις προσπάθειες που καταβάλεις.